Και οι πολιτικές και οι οικονομικές λοιπόν μεταρρυθμίσεις είναι προϋπόθεση για ένα καλό μέλλον για την Ουκρανία που θα είναι προς το καλύτερο συμφέρον των πολιτών της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλεάν <clears throat> για τους πράσινους Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία η κυρία Χάμς για δύο και μισά